Επομένω, επικυρώνονται οι εντολέ των δύο οι βουλευτικές των δύο αυτών συναδέλφων. Τώρα περνούμε στις, ε, στα νομοθετήματα που εξετάζονται με τη διαδικασία της συναπόφασης. Θα σας ενημερώσω ότι συζητήσαμε στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την τελευταία εβδομάδα βάσει του άρθρου 74 ε, του κανονισμού. Πρόκειται για πράξεις οι οποίες θα δημοσιευθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.